Ε, θα υπάρξουν κάποιες οδηγίες αν θέλετε για την σημερινή συνεδρία. και αυτό αφορά τα μέλη μας βέβαια. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Μετά από την ακρόση που έγινε χθε, το μόνο θέμα που έχουμε σήμερα είναι η ψηφοφορία ε, του ελεγκτή και του βοηθού ελεγκτή. Θα υπάρχει διευμηνία σε 20 γλώσσες αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την δανική Ε, θα, ναι μεν μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και χθε έλαβα υπόψη την παρατήρηση της κυρία Ίντβελτ σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής την οποία ακολουθήσαμε. Κοιτάξτε, εγώ ως πρόεδρος και ζητά πάλι ησυχία Δεν ξέρω αν όλα τα σχόλια του Επιτρόπου ήσαν πλήρως κατανοητά. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία παρά το ότι η διαδικασία μπορεί να είχε κάποια προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Και αν υπάρχουν σχόλια από πλευρά των συντονιστών μπορούν να τα εκφράσουν τώρα. Αλλά εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στις ψηφοφορίες γιατί η ενημέρωση στην οποία είχαμε στη διάθεσή μας ήταν επαρκής. Γι' αυτό παρακαλώ θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την παρατήρηση της κυρίας Ιντβελ Χέλτ. Ζόφι, θες να κάνεις ε, μια παρατήρηση. Κοιτάξτε, τουλάχιστον να μας δοθούν κάποιες διευκρινήσεις εκ των υστέρων έστω. Κοιτάξτε, σίγουρα η επιστολή δεν ήταν επαρκής απάντηση Γι' αυτό αν έχετε κάποια στοιχεία επιπλέον να μας δώσετε μπορείτε να το κάνετε τώρα. Ε, Κλοντ, ε, έχω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε ε, τι σημασία έχει αυτό το οποίο εμείς αποφασίζουμε σε σχέση δηλαδή με το, τις αποφάσεις του Συμβουλίου κατά πόσο έχει βαρύτητα η δική μας απόφαση πριν ψηφίσουμε, καλό θα ήταν να μας δοθούν αυτές οι διευκρινήσεις. Εγώ δεν ε, ε, ε, θεωρώ ξεκάθαρο το τι ακριβώς κάνουμε σε αυτή την ψηφοφορία. Okay, Cornelia, I'm going to um, read out a set of... Um, λοιπόν, θα σας διαβάσω κάποιες οδηγίες εισαγωγικά και ελπίζω αυτό να σας καλύψει. Αν έχετε κάποιες απορίες μετά από αυτά τα οποία θα πω να αντιστέσετε. Να ξεκινήσω με κάποιες από τις λεπτομέρειες τις οποίες χρειάζεστε. Η διαδικασία ακολουθεί το άρθρο 42 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφέρεται στην κοινή γνώμη και συμφωνία για τον ελεγκτή και τον βοηθό ελεγκτή για μία περίοδο 5 ετών. Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν εμπειρίες και εμπειρογνωμοσύνη απαιτούμενοι από τις ε, ε, ενέργειες στις οποίες θα κληθούν να λάβουν μέρος. Να πω στους συναδέλφους που δεν ήταν χθε ίσως στην ακρόαση ότι αυτά, τα, αυτές οι λεπτομέρειες είναι απαραίτητες και να πω ότι κάθε υποψήφιος ανέφερε ότι θα δεχθεί τις ε, θέσεις αυτές τις οποίες έχουμε σαν Επιτροπή και όλοι εκτός από έναν τις εδέχθησαν. Υπάρχουν πέντε λοιπόν υποψήφοι και τέσσερις για την θέση του βοηθού ελεγκτή. Ο κύριος Πάντοβα δεν είναι υποψήφιος, είπε ότι δεν ήθελε ε, να είναι υποψήφιος βοηθός ελεγκτής. Η ψηφοφορία θα γίνει ως εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 181 και με το άρθρο 182 η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική και μυστική. Χρειάζεται δηλαδή η κάρτα σας, η ηλεκτρονική. Ετοιμάστε την παρακαλώ. Πρώτα θα καθορίσουμε την σειρά προτίμησης για την θέση του ελεγκτή. Θα ψηφίσουμε για τον καθένα από τους πέντε υποψηφίους και μετά θα γίνει μια δεύτερη ψήφος για να φτιάξουμε ένα κατάλογο προτιμήσεων για τον βοηθό ελεγκτή. Δεν έχει την κάρτα της η συνάδελφος και θα θέλαμε να μπορέσει να ψηφίσει. Οκ, okay, κάποιος θα της δώσει όμως μια άλλη κάρτα. θα πρέπει σαν συντονίστρια να γνωρίζεις ότι δεν πρέπει να μου κόβεις τη φόρα. Αυτό μου δημιουργεί θέματα. Νόμιζα ότι το είχαμε μάθει αυτό. Λοιπόν σας έλεγα ότι θα ακολουθήσει Οι πράσινοι γενικά συζητούν μεταξύ τους. Θα γίνει μια δεύτερη ψήφος για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας για τον βοηθό ελεγκτή. Έχουμε τέσσερις υποψηφίους και θα ψηφίσουμε για τους τέσσερις. Πέντε λοιπόν υποψήφοι στη θέση του ελεγκτή και τέσσερις στη θέση του βοηθού ελεγκτή. Θα λάβουμε υπόψη μας μόνο τις θετικές ψήφους μπορείτε να ψηφίσετε μόνο θετικά, αν θέλετε. Δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, δεν μπορείτε να καταψηφίσετε. Το πράσινο είναι στα αριστερά σας. Προλαβαίνω την ερώτηση. Το πράσινο είναι αριστερά λοιπόν. Δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ψήφο σας εκ των υστέρων. Λοιπόν, αριστερά σας το πράσινο κουμπί. Το κόκκινο ε, είναι αρνητικό. Αν θέλετε να καταψηφίσετε τότε απλά δεν ψηφίζετε. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα σήμερα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας κατάλογος των υποψηφίων ανάλογα με την λίστα που θα δημιουργηθεί θα ξεκινήσουμε για τον ελεγκτή. Οι ψήφοι θα καταγραφούν από την γραμματεία και από μένα και το ίδιο θα κάνουμε και με τον κατάλογο που θα διαμορφωθεί μετά την ψηφοφορία για τον βοηθό ελεγκτή. Εγώ θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα μόνο μετά το τέλος όλων των ψηφοφοριών. Καμία πληροφορία πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γι' αυτό μην ζητάτε παρακαλώ πληροφορίες για συγκεκριμένους υποψηφίους να πω ότι όπως είπαμε χθε θα ψηφίσουμε με τη σειρά που παρουσιάστηκαν οι υποψήφοι χθε το απόγευμα. Για τη θέση του ελεγκτή λοιπόν, πέντε υποψήφοι όπως είπα, όταν ξεκινήσουμε αν οι πολιτικές δυνάμεις εκπροσωπούνται πλήρως πριν την ψηφοφορία θα το ελέγξουμε αυτό και θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ψηφίστε όπως θέλετε να ψηφίσετε και θα δούμε ε, πόσοι ψηφίζουν από κάθε πολιτική ομάδα. Θέλετε να υπάρξει μία ψήφος ελέγχου δοκιμαστική πρώτα. Ναι, καλό είναι, λένε κάποιοι από εσά να υπάρξει μια δοκιμαστική ψήφος. Λοιπόν, δοκιμαστική ψήφος. Ψηφίστε παρακαλώ θετικά για κάτι. Ψηφίστε όλοι θετικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα επιπλέον μέλος ε, ε, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή ένας επιπλέον δεν μπορεί να ψηφίσει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες έχουν τον σωστό αριθμό ψήφων. Γι' αυτό λοιπόν οι συνάδελφοι του ΕΛΚ θα πρέπει να εξαιρέσουν ένα συνάδελφο από την ψηφοφορία και παρακαλώ να μην αλλάξετε, κρατήστε τις θέσεις σας και ψηφίστε στη θέση στην οποία βρίσκεστε. Εντάξει, συμφωνείτε. Διαδικαστικά δύο συνάδελφοι. Κοιτάξτε, μιλάμε για αυτούς που θα προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά αν εμείς ε, δεν ψηφίσουμε γιατί το κόκκινο δεν δουλεύει όπως είπατε, αυτοί που δεν θέλουν ε, να ψηφίσουν θα φανεί ε, ότι δεν ψηφίζουν. Αν κάποιος ψηφίσει ε, το πράσινο, πατήσει το πράσινο φαίνεται. Άμα δεν ψηφίσει επίσης δεν ανάβει το φωτάκι, οπότε γνωρίζει ο άλλος ότι δεν έχεις ψηφίσει. Και αυτό δεν είναι σωστό, δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της διαδικασίας. Η ψηφοφορία θα πρέπει να είναι μυστική, δεν πρέπει να φαίνεται αν κάποιος δεν ψηφίζει. Κοιτάξτε, ε, Νομίζω ότι πρέπει να επιτρέψουμε να πατάει κανείς το πράσινο κουμπί ή το κόκκινο κουμπί γιατί αλλιώς η ψηφοφορία δεν είναι μυστική λέει ο κ. Κοέλιο. Κοιτάξτε έτσι και αλλιώς το πράσινο φαίνεται μπλε λέει ο πρόεδρος. Κατανοώ αυτό το οποίο λέτε. Ε, λέτε ότι τη στιγμή που ψηφίζεται κάποιος μπορεί να δει το τι ψηφίζεται. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Παρακαλώ λίγη ησυχία συνάδελφοι. Uh, look, I think that's it. Colleagues, can, if you stay quiet for a moment, I'm just going to respond to. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπατε. Ε, είναι λογική η πρόταση την οποία κάνατε, θετική πρόταση αν κάποιος παρακολουθεί την ψηφοφορία και βλέπει τι κάνει ο άλλος αυτό δεν είναι σωστό γιατί είναι ευαίσθητη η ψηφοφορία οπότε σας προτείνω αν θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε και κόκκινο δεν είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν ψηφίζετε το πράσινο αλλά μπορείτε να ψηφίσετε και κόκκινο αν αυτό διευκολύνει την ψηφοφορία λοιπόν είναι μια επιπλέον λεπτομέρεια που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα Λοιπόν, αν πατήσετε κόκκινο, πάντα θα φαίνεται ε, ότι ψηφίζετε, αλλά δεν θα ξέρει ο άλλος τι ψηφίσατε. Ακόμα και αν δεν ψηφίζετε, γιατί είπαμε μόνο το πράσινο μετράει. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, λέει η κυρία Σίπελ. Όπως είπαμε και στον πρώτο γύρο, μόνο οι θετικές ψήφοι είναι εφικτοί. Οπότε αν θέλει κανείς να ψηφίσει για έναν και για δύο δεν το κάνει για τους υπόλοιπους. Αλλά για να υπάρχει φωτάκι πάντα ε, ε πατώντας τα κουμπί έτσι και αλλιώς το φωτάκι θα μένει ανοιχτό οπότε οι άλλοι δεν θα καταλαβαίνουν τι ψηφίζουμε. Κοιτάξτε είπατε το ίδιο που είπε ο κύριος Κοέλιο. Λοιπόν, πάντα χρειάζεται κάποιος από αυτή την ομάδα για να σε επιβεβαιώνει τι θα κάνουμε. Και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα των σοσιαλιστών, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ας περάσουμε στην ψηφοφορία, συνάδελφοι. Λοιπόν, πίστευα ότι θα τελειώναμε γρήγορα, αλλά δεν φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Περνάμε λοιπόν πρώτα, συνάδελφοι, Λοιπόν, δεν έχει και τρομερό ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε. Ο πρώτος υποψήφιος ελεγκτής είναι ο κύριος Βιβορόφσκι. Βιεβιεβορόφσκι. Άρχεται η ψηφοφορία για τον κύριο Βιεβιεβορόφσκι. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Okay. Okay, Mr. Engel, did you have a disturbing point of order right in the middle of votes? Κύριε Έγγελ, μας ενοχλεί το διαδικαστικό σας. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Έγγελ, αν κατάλαβα καλά, η προστασία των δεδομένων Ε, δεν οδηγεί στο να δουλεύει μόνο το ένα από τα τρία κουμπιά. Στην περίπτωση τη δική μου μόνο ένα από τα τρία κουμπιά δούλεψε. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ψήφισα λάθος. Γιατί δεν μπορώ να ανακαλέσω την ψήφο μου. Και η ψήφος την οποία θα ήθελα ε, να δείξω ε, δεν, είναι, δεν στάθηκε δυνατό να το κάνω. Okay, change, change your seat anyway, and we'll look into that for... Κοιτάξτε, αλλάξτε τη θέση σας και θα το λάβουμε υπόψη μας. Κοιτάξτε, ας μην καθυστερήσουμε συναδέλφοι. Αλλάξτε θέση κύριε Έγγελ. Though, because we're going on to the next vote. Insert your card quickly because I'm moving on to the next vote. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα ξαναγίνει δυστυχώς η ψηφοφορία. Δεν θέλω να σας να ρίξω κανέναν, αλλά για λόγους ακρίβειας θα ξαναγίνει η ψηφοφορία για τον κύριο Βιβορόφσκι, για τη θέση του ελεγκτή. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε για τον κύριο Βιβορόφσκι. Scommetto che quando usciremo da questa parte dove andremo. The vote is closed. Okay, colleagues. Πέρασε τη ψηφοφορία. Συνάδελφοι, για την κυρία Μπιόντι τώρα η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την κυρία Μπιόντι. Πέραση της ψηφοφορίας. E Τώρα για τον κύριο Μπουταρέλη για τη θέση του επόπτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι έγινε. Για τον κύριο Μπουταρέλη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει μία ψήφο παραπάνω. Ωραία, πάει. Έφυγε η παραπάνω ψήφος, πέρασε η ψηφοφορία. Τώρα για, την κυρία Λενουάχ, για τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και για τον κύριο Πάντοβα, άρχεται η ψηφοφορία για τη θέση του Επόπτη και πάλι. Πέρας της ψηφοφορίας. Τώρα για τη θέση του αναπληρωτή επόπτη ψηφίζουμε για τον κύριο Βιβερόφσκι. Άρχεται η ψηφοφορία για τον κύριο Βιβερόφσκι. Πέρας της ψηφοφορίας. Για την κυρία Μπιόντι, άρχεται η ψηφοφορία για τη θέση του αναπληρωτή επόπτη ε, ε, Προστασία Δεδομένων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Για τον κύριο Μπουταρέλη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψυχοφορίας. Και για την κυρία Λενουά άρχεται η ψηφοφορία για τη θέση του αναπληρωτή επόπτη. Πέρας της Colleagues, I'm just going to verify this with the Secretary. Πριν σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα θα τα ελέγξουμε με τον γραμματέα. Ε, αφήστε με λοιπόν μισό λεπτάκι. Ε, τώρα αγαπητοί συνάδελφοι θα σας ανακοινώσω τη σειρά και τον αριθμό ψήφων για κάθε θέση. Καταρχήν για τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη τα αποτελέσματα έχουν ω εξή. Πρώτη προτίμηση δίνεται στον κύριο Τζοβάνι Μπουταρέλη, 34 ψήφοι. Δεύτερη, 21 ψήφοι για τον κύριο Γιάν Πάντοβα. Τρίτη προτίμηση για τον κύριο Βιβερόφσκι, 10 ψήφοι. Τέταρτη η κυρία Λενουάχ με 4 ψήφου. Και πέμπτη η κυρία Μπιόντι με μία ψήφο. Για τη θέση του αναπληρωτή επόπτη ε, προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Βιβερόφσκι πρώτος με 53 ψήφους, ο κύριος Τζοβάνι Μπουταρέλη δεύτερος με 9 ψήφους, η κυρία Νοέλ Λενουάρ τρίτη με 3 ψήφους, και τέταρτη κυρία Μπιόντι με δύο ψήφους. Θα στείλω μια επιστολή στον Πρόεδρο για να τον ενημερώσω για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Θα είναι καθήκον μου να είμαι σε επαφή με την Προεδρία του Συμβουλίου για να καταλήξουμε στην κοινή συμφωνία που προβλέπετε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 45 του 2001. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.